President. και αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η επίσημη πανηγυρική συνεδρίαση που τελείται επί τη δεκαετή επαιτίο της, ε, ε, του, του Κοινού Ευρωπαϊκού Νομίσματος του Ευρώ.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 Herr Premierminister und Präsident der Κύριε Πρωθυπουργέ ε, Jean-Claude Juncker, κύριε Πρόεδρε ε, Giscard d'Estaing, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κύριε Τρισέ, κύριε Επίτροπε, κύριε Αλμούνια, αγαπητοί ε, Πρόεδρε της Επιτροπής Νομισματικών Θεμάτων, κύριε Μπερές, κυρίες και κύριοι, την 1η Ιανουαρίου 2009 το κοινό μας ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ, γίνεται 10 ετών. Εορτάζουμε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία από τις πιο σημαντικές ιστορικές αποφάσεις που έλαβε στην ιστορία της Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημιουργία του ευρώ μέσα στα πλαίσια μιας οικονομικής ένωσης που γινόταν όλο και πιο στενή ήταν μια λογική εξέλιξη για την διευκόλυνση του εμπορίου και για την εναρμόνιση των πολιτικών. Προ λοιπόν η, τα εθνικά νομίσματα 11 χωρών μελών αντικατάστηκαν από ένα κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Είχαν εκφραστεί πολλές επιφυλάξεις τότε σχετικά με την επιτυχία του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Η εισαγωγή του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος απίτησε αποφασιστικότητα και θάρρος. Μία δεκαετία μετά διαπιστώνουμε ότι το ευρώ απολαμβάνει την εμπιστοσύνη ε, του κοινού όπως και τότε τα ε, ξεχωριστά ευρωπαϊκά νομίσματα. Η Ευρωζώνη έχει γίνει μια ζώνη μεγάλης οικονομικής σταθερότητας. Εν ώψη του βάρους της και του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου είναι εσωτερικό εμπόριο, η Ευρωζώνη είναι ισχυρότερη από το σύνολο των χωρών μελών για να αντιμετωπίσει τις διακυμάνσεις της παγκόσμιας οικονομίας. Τα τελευταία, ε, τους τελευταίους μάλιστα μήνες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το ευρώ αποδεικνύεται σημαντικός παράγοντας σταθερότητας. Το κοινό νόμισμα ε, μας προστάτευσε από τις ε, σημαντικότερες διακυμάνσεις της βαρύτερης κρίσης που έχει σημειωθεί στην παγκόσμια οικονομία από τη δεκαετία του 1930 χωρίς το σύστημα αυτό. Χωρίς το σύστημα των, ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως το φθινόπωρο του 2008 θα ήταν κατά πολύ χειρότερη. Η Ισλανδία για παράδειγμα, μια χώρα η οποία πλήγει βαρύτατα από την οικονομική κρίση. Μια ε, παρόμοια περίπτωση θα μπορούσε να είναι η Ιρλανδία που όμως ε, διασώθη λόγω του ότι ανήκει στην Ευρωζώνη. Είναι λοιπόν ανεπίστρεπτο το βήμα αυτό προς την κατεύθυνση μιας ε, ε, στενότερης οικονομικής συνεργασίας. Γιατί σημαίνει μια ένωση με ένα κοινό προορισμό. Όπως τα μέλη μιας οικογένειας, όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνομιλούν και συναποφασίζουν για το ποια είναι η ε, καλύτερη οδό για την εξασφάλιση των συμφερόντων κάθε μιας χώρα ξεχωριστά και όλων μαζί. Όμω δεν είναι μόνο οι οικονομικέ οι επιπτώσει τη χρήση του ευρώ, είναι και σαφέ το μήνυμα το οποίο δίνει ότι η Οικονομική Ένωση είναι σε θέση να λάβει μακροπρόθεσμες αποφάσεις για να εξασφαλίσει το κοινό μέλλον εν ευημερία. Σήμερα το κοινό νόμισμα θεωρείται από πολλούς πολίτες των χωρών της Ευρωζώνης ως ένα από τα πιο θετικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να παραμείνει αυτό έτσι και στο μέλλον, οφείλουμε να εργαστούμε έτσι περαιτέρω για την σταθερότητα του κοινού μας ευρωπαϊκού νομίσματος. Μόνο έτσι το ευρώ θα παραμείνει και στο μέλλον παράγοντας σταθερότητας και μια άγκυρα για το σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ταραγμένα νερά της παγκόσμιας οικονομίας. Προδεκαετίες λοιπόν εισήγαν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προ λίγων μερών η ε, Σλοβακία εντάχθηκε ως 16η χώρα στην Ευρωζώνη. Ελπίζω στις επόμενες επαιτίους του ευρώ να μπορέσουμε να υποδεχθούμε ή να έχουμε υποδεχθεί στο μεταξύ και άλλα μέλη στην ζώνη ευρώ. Μια τέτοια βαθμιδών επέκταση απαιτεί και απαιτείται για την σταθερότητα της Ευρωζώνης και ιδίως στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσφέρει την δυνατότητα ε, διασφάλισης ενός ειρηνικού μέλλοντος. Σήμερα είναι μαζί μας ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Βαλερίου Ζισκάρντεστα. Του απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό και μαζί με τον Χέλμουντ Σμιτ τον ε, Πιέρ Βέρνερ του Λουξεμβούργου είναι μεταξύ των αρχιτεκτόνων του κοινού νομίσματος. Καλώς ήρθατε μεταξύ μας Βαλερή Καντεστάν. Θα συμφωνήσω με τα λόγια του Helmut Kohl, ο οποίος μαζί με τον Φρανσό Μιτεράν, τον Ζακ Ντελόρ και άλλες προσωπικότητες και τον Ζακ Σαντέρ που τον είδαμε προηγουμένως στο βίντεο. Είναι μεταξύ των προσώπων εκείνων που συνέβαλαν στην τελική εισαγωγή του ευρώ. Ο Helmut Kohl έλεγε λοιπόν το 1998 ότι ένα νόμισμα είναι βεβαίω ένα μέσον πληρωμής, αλλά είναι και πολύ περισσότερα πράγματα από ένα μέσον πληρωμής. Ε, συναποτελεί και την ταυτότητα και ένα σημάδι σταθερότητας. εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλη την ευφυΐα, όλη τη δημιουργικότητα της Ευρωπαϊκής Επίρου ότι περισσότερα από, 500 περισσότερα από 200 ε, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν το κοινό νόμισμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, στο όνομα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους τους αρχιτέκτονες του ευρώ να ευχηθώ ιδίω στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πρόσωπο του σημερινού της Προέδρου Jean-Claude Trichet αλλά και θυμούμενος τον πρώιμα αποβιώσαντα Βίλεμ Ντάιζενμπεκ, τον προκάτοχό του. Σας ευχαριστώ λοιπόν ειλικρινά και από βάθος καρδίας. Είναι σημαντικότατος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι ευχαριστίες μου ανήκουν και στον Αλεξάνδρου Λαμφαλουσί, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου. Τον συναντήσαμε χθε και συμμετέχει και σε συμπόσιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η αρμόδια επιτροπή του, η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή υπό την προεδρία του τότε πρόεδρου της Κάλφον Βόγκαου και με την ε, διάδοχό του Κρίστα Ράντζιο Πλάτ κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες που ήταν αποφασιστικές για την ε, πρόθεση του κοινού νομίσματος. Το ίδιο ισχύει και για την σημερινή Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή υπό την ηγεσία της Περβάνς Μπερές η οποία μάλιστα είχε και την ιδέα της σημερινής εορταστικής εκδηλώσεως. Προδεκαετίας οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες και η Ευρωομάδα άρχισαν τακτικές επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η καλή αυτή συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αποδώσει. Απευθύνω λοιπόν χαιρετισμό στον κύριο Ζαν Κλοντ Juncker που είναι πρόεδρος της ομάδας της Ζώνης Ευρώ καθώς και τον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας και πάλι κύριο Ζαν Κλοντ Τρισέ. Για την δέκατη επέτειο, για τα δέκατα γενέθλια του ευρώ ευχόμαστε στο κοινό μας νόμισμα πολλά επιτυχή χρόνια για την εξασφάλιση ε, του κοινού μέλλοντος της Ευρωπαϊκής μας Επίρου. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να είναι ακόμη πολύ αριθμότεροι συνάδελφοι, αλλά τουλάχιστον εσείς είστε εδώ και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο τώρα στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ. Jean-Claude Trichet. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά για μένα που συμμετέχω σε αυτήν την τελετή που γιορτάζει μια από τις, τα βασικά επιτεύγματα της Ευρώπης που είναι ο Ευρώ ένας από τους ιδρυτής της Ενωμένης Ευρώπης, είπε ότι όταν μια ιδέα ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα της εποχής πάβει να ανήκει σε αυτούς που την επινόησαν ε, και ανήκει περισσότερο σε αυτούς που την έχουν αναλάβει. Υπάρχουν σκόπιμες στιγμές, εύστοχες που κάποιος θα πρέπει να περιμένει. Αυτό το ευρώ ήταν μια ιδέα που συμμεριζόντουσαν λίγοι, ενώ οι άλλοι, οι περισσότεροι πίστευαν ότι θα ήταν αποτυχία. Σήμερα το ενίο νόμισμα είναι μια πραγματικότητα για 329 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Μια μέρα η δημιουργία του ευρώ θα θεωρηθεί ως αποφασιστική ε, καμπή στο δρόμο ε, μιας ένωσης που ε, φέρνει όλο και πιο κοντά τους ευρωπαϊκούς λαούς. Είδαμε τους ιδρυτές, τον Ρόμπερ Σουμάν, τον Βαλστάιν, Αλσίντε Γκάσπερι, Πιερ Βερνέρ, Σίκο Μάντσχολτ, Πολόν Σπάκα. Σκέφτομαι επίσης τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που υπήρξαν ε, πεπισμένοι Ευρωπαίοι, θαραλέοι, υπέρ της ιδέας της Ευρώπης και που τους αντιπροσωπεύει εδώ ο πρόεδρος Βαλερή Γίσκαρδεστά. Χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε το ευρώ από την εισαγωγή του ευρώ οι συμπολίτε μας έχουν ένα επίπεδο σταθερότητας τιμών που μόνο μέχρι τότε είχαν ορισμένες χώρες. Είναι ένα πλεονέκτημα για το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών, προστατεύουν τα εισοδήματά τους, την αποταμίευσή τους, μειώνουν το κόστος χρηματοδότησης, προστατεύουν την ευημερία μακροπρόθεσμα. Είναι ένα παράγον δυναμισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία, βελτίωσε την διαφάνεια των τιμών, ευνόησε της ανταλλαγής και την ολοκλήρωση την οικονομική και την ε, χρηματοοικονομική. Βλέπουμε τελευταία στα γερμανικά ακόμα ένα πλεονέκτημα του ευρώ. Η χρηματοπιστωτική κρίση δείχνει ότι σε ταραγμένους καιρούς είναι καλύτερο να ε, είναι κανείς ένα πλοίο μεγαλύτερο και ασφαλέστερο ε, παρά σε ένα μικρό σκάφος. Λιγότερο αξιόπλο. Εάν στην Ευρώπη δεν είχαμε ε, το κοινό νόμισμα δεν θα μπορούσαμε ε, να αποφασίσουμε τόσο γρήγορα και τόσο σωστά. Θα είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τις εθνικές οικονομίες από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Άραγε νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι ε, στις αντιδράσεις των κοινοβουλίων, των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών στην Ευρώπη. Από κοινού δείξαμε ότι η Ευρώπη ακόμα και στις πιο δύσκολες περιστάσεις είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις. Στα αγγλικά τώρα. Ε, η ιστορική επιτυχία του ευρώ δεν οφείλεται μόνο στη διορατικότητα και ε, στην επιμονή των ηγετών αλλά και ε, στην καλή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αρχικό στάδιο έπαιξε ρόλο πρωτοπόρο και κρίσιμο. Ήταν το πρώτο θεσμικό όργανο που έκανε πρόταση ήδη από το 1962 και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάντα υπήρχε διάλογος μόνιμος και γόνιμος. Πάνω από 50 ακροάσεις είχαμε τα μέλη του ε, Εκτελεστικού Συμβουλίου της ε, Τράπεζας πριν ε, καταλήξουν το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Ο διάλογος Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι πάρα πολύ σημαντικός για όρους δοσίας για να ε, εξηγεί ε, στο ευρύ κοινό η τράπεζα τις αποφάσεις και τις ενέργειές της μέσω των ερετών προσώπων του ε, Ευρωπαϊκού Τρία ήταν, τρεις ήταν συγγνώμη, μεγάλες δοκιμασίες για το ευρώ. μια υγιής κεντρική τράπεζα ίδρυσή της, δηλαδή η δημιουργία ενός σταθερού νομίσματος που να εμπνέει εμπιστοσύνη και σταθερότητα. Σιγά σιγά ξεπεράσαμε αυτές τις προκλήσεις και είναι γερά εδρεωμένο σήμερα το ευρώ και έχει έρθει η ώρα ε, για τους εορτασμούς πανηγυρικούς. Σας είπα ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Χωρίς σημαίνει ότι θα πρέπει να εφησυχάζουμε. Έχουμε ξεπεράσει κάποιες προκλήσεις αλλά οι νέες καταφθάνουν ε, και η επιτυχία του ευρώ θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα τις αντιμετωπίσουμε. Να σας πω ποιες είναι αυτές τρεις. Η χρηματοπιστωτική κρίση. Είδαμε ότι το ε, παγκόσμιο σύστημα έχει ε, κλονιστεί στα θεμέλια του, προσπαθούμε να ε, ξανασχεδιάσουμε το θεσμικό και το κανονιστικό πλαίσιο. Δεύτερον, η νομισματική ένωση. Ε, η πυγμή και η σταθερότητα του νομίσματος βασίζεται σε δύο πυλώνες νομισματική σταθερότητα, σταθερότητα των τιμών και στη συνέχεια υγιής οικονομική πολιτική που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό στα χέρια της Ευρωβάδας, κύριε Γιούγκερ θα πρέπει ε, αξιόπιστα ε, και ε, σταθερά, να εφαρμόζεται το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη για να είναι πιο ενεργέ οι οικονομίε, πιο δυναμικέ και να μην έχουμε μεγάλε ανταγωνιστικέ αποκλήσει στην Ευρωζώνη. Τρίτον, η διεύρυνση. Όταν ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια το ευρώ, ήμασταν 11 χώρε. Σήμερα είμαστε 16 χώρε στην Ευρωζώνη και αυτό λέει πολλά για το ιστορικό αυτό εγχείρημα. η σωστή και καλή διεύρυνση είναι πάντα πρόκληση για μας, απαιτητική, ε, που μας εμπνέει όμως και όλους. Αυτό το λέω και εξ ονόματος της ηγεσία της τράπεζας. Το ευρώ είναι ιστορικό επίτευγμα και αυτό που σήμερα έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η ευθύνη μας για το μέλλον. Έχουμε νέες προκλήσεις ε, που αναδύονται και αν τις ε, αντιμετωπίσουμε με τόλμη και με παρησία ε, τίποτα δεν θα μας εμποδίσει να ε, προωθήσουμε τις ιδέες του Ζαμονέ στο μονοπάτι και στην οδό της ε, σταθερότητας και της ευημερίας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στα γαλλικά. Στα γαλλικά και ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για την ομιλία σας και τη μεγάλη σας προσήλωση και δέσμευση. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους πρώην Προέδρους του Κοινοβουλίου, ε, Χωσέ Μαρία Χιρόμπλες, Χιλτελγκάδο, Νικόλ Φοντέ, Ρίκε Μπαρόν Κρέσπο και Κλάους Χένς. Ε, χαίρομαι που βρίσκεστε σήμερα ενώπιόν μας. Παρακαλώ τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Ευρωομάδας, Ζανκλότ Γιούγκερ, να λάβει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Κατά τη διάρκεια των 50 τελευταίων ετών η Ευρώπη συχνά απέδειξε την ικανότητά της ε, να εκφράζει μεγάλες φιλοδοξίες και την ικανότητά της ε, να αναπτύσσει το απαιτούμενο πνεύμα και την απαιτούμενη βούληση και αποφασιστικότητα που χρειάζονται ε, για την συνεπή υλοποίηση των φιλοδοξιών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια είναι το καλύτερο παράδειγμα αυτής της βούλησης όπως η εσωτερική αγορά, όπως η διεύρυνση, δηλαδή ε, η προσέγγιση, η γεωγραφική ε, στην ευρωπαϊκή ιστορία και όπως ε, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση της οποίας γιορτάζουμε σήμερα τη δεκάτη επέτειο. Ο δρόμος που οδήγησε στην δημιουργία της ΟΝΕ και στην εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος ήταν μακρύς δρόμος και η γέννηση της ΟΝΕ με την αρχική όθηση της εισήγησης του 70 του Βέρνερ το αποδεικνύει μια γέννηση που πέρασε από το φίδι το νομισματικό, από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, την δημιουργία του ΕΚΙΟΥ το 1979, το πρόγραμμα Delors του 89, τη συνθήκη του Μάστριχ του 1992, όπως επίσης με το όχι το δανεικό και το ναι το γαλλικό που την εποχή εκείνη λέχθηκε μικρό χωρίς να ξεχάσουμε την ε, κρίση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος του 1993. Όλο αυτό το ταξίδι, όλο αυτός ο περίπλους δεν έγινε χωρίς ε, δυσκολίες ή χωρίς ε, συγκρούσεις. Πολλοί ήταν την εποχή αυτή που ήταν κατά του ενιαίου νομίσματος, είτε στους πολιτικούς κύκλους, είτε στους ακαδημαϊκούς, χωρίς ε, να ξεχάσουμε ένα σημαντικό αριθμό κεντρικών τραπεζιτών που εκτιμούσαν ότι ο ναι δεν μπορούσε να γίνει ή δεν έπρεπε να γίνει και αν έπρεπε να πραγματοποιηθεί παρόλα αυτά το ενιαίο νόμισμα Φίνε θα ήταν ένα ασθενές νόμισμα χωρίς επαύριο. Πρέπει λοιπόν να υποφεληθούμε από την δεκάτη επέτειο αυτού του γεγονότος, του σημαντικού της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης για να αποτίσουμε φόρο τιμή σε αυτούς που δημιούργησαν το, το ευρώ, τον Χερμουτ Κόλ, Βέρνερ, Φρανσουά Μιτερό, Ζακ Ντολόρ, Βαλερί Καρδεστάν και άλλους. Θα ήθελα εδώ άλλη μια φορά να χαιρετήσω, να αποτίσω φόρο τιμή στο όραμά τους, στην αποφασιστικότητά τους, στη δέσμευσή τους την αδιάλειπτη. Πολλοί άλλοι τους συνόδευσαν ε, όλοι αυτοί δεν θα μπορούσαν να φανταστούν την τόσο ταχεία επιτυχία ε, του πολιτικού τους ε, σχεδίου. Από την 1η Ιανουαρίου έχουμε 16 κράτη-μέλη στην ΟΝΕ και έχουμε περίπου 330 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που έχουν το ευρώ ως επίσημο νόμισμα. Είναι το πιο, η πιο απτή απόδειξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που αναγνωρίζεται παντού στον κόσμο. Το ευρώ είναι αν θέλετε ένα σπυρίνα σταθερότητας και προστατεύει τους πολίτες από τις δυσμενείς επιπτώσεις οικονομικής κρίσης. Μετά από δέκα χρόνια πρέπει να διαπιστώσουμε ότι το ευρώ είναι ανδιαμφισβήτητη επιτυχία. Οι επέτειοι αξίζουν μόνο αν αποτελούν γέφυρες προς το μέλλον και πρέπει επίσης να διαπιστώσουμε ότι παρά την συλλογική επιοίκεια και το ότι συνέχεια αυτό συγχαιρόμαστε, πρέπει να έχουμε ε, μια, πολλά να κάνουμε για την συνεκτικότητα και την συνοχή του ευρωπαϊκού χώρου. Το 2009 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τις ευρωχώρες και για τους ευρωπαίους πολίτες και πολλές θα είναι οι προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τόσο στο εσωτερικό όσο και εκτός. Στο εσωτερικό οι κυβερνήσεις ε, του ευρωχώρου θα πρέπει να δράσουν μαζί για να συγκρατήσουν ε, τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης ε, και να επενδύσουν στις βάσεις της διαφορετικής οικονομίας για να δημιουργήσουν μια γέφυρα για μετά την κρίση. Οι εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν εξαιρετικά μέτρα. Έκτακτα μέτρα, έκτακτες περιστάσεις, έκτακτα μέτρα Βεβαίω, όλα αυτά τα οποία έχουμε δεν δημιουργήθηκαν από το τίποτα. Οι οικονομίε μα είναι καλύτερα προστατευμένε από τι αρνητικέ συνέπειες διότι το ότι ανήκουμε στο ευρώ είναι ένα σήμα ποιότητας που δείχνει ότι έχουμε την ικανότητα να έχουμε μακροοικονομικές πολιτικές προσεκτικές που είναι προσαρτολισμένες προς την διαιώνιση της οικονομικής μεγέθυνσης και την ευημερία των πολιτών διότι όλα αυτά σχετίζονται με την αξιοπιστία μας να υλοποιήσουμε αυτές τις πολιτικές. Αυτή η αξιοπιστία είναι ε, το θεμέλιο των πλεονεκτημάτων της ΟΝΕ και θα πρέπει ε, να την χρησιμοποιήσουμε για να μπορούμε να επωφεληθούμε πλήρως από τα πλεονεκτήματα του ενιαίου νομίσματος. Ε, στο εξωτερικό θα πρέπει να επωφεληθούμε διότι υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στην σημερινή κρίση με τα αίτια στις Ηνωμένες Πολιτείες και την εμμονή ε, των ε, ανοσορροπιών των παγκοσμίω. Η έλλειψη διαφάνειας και ακαιρεότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα ε, μετά υπήρξε καταλήτης της κρίσης. Η αποκατάσταση της σταθερότητας της χρηματοπιστωτικής οικονομίας και της πραγματικής οικονομίας απαιτεί εις βάθος μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και επίσης την εξάλληψη των σημαντικών ανισορροπιών στο μείγμα ανάμεσα στην συνολική κατανάλωση και στην συνολική αποτέμιευση. Αυτό απαιτεί την συνεργασία μεταξύ των μεγάλων οικονομιών Αμερικής, Ασίας και Ευρώπης. Παρά στις σημαντικές προόδους, η εκπροσώπηση διεθνής του ευρώ είναι συχνά κατατεμαχισμένη και εθνικά συμφέροντα επικρατούν πολύ συχνά πάνω στα κοινά συμφέροντα και εμποδίζουν τον χώρο του ευρώ να αναλάβει πλήρως τις πολιτικές ευθύνες που αντιστοιχούν στο οικονομικό βάρος της Ευρώπης και για να υπάρξουν τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη στα οποία προσδοκούμε. Η είναι ένα σχέδιο ε, ε, οικονομικό αλλά πρώτα απ' όλα πολιτικό. Πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε ε, την δεύτερη δεκαετία του ευρώ για να τελειοποιήσουμε την ΟΝΕ ενισχύοντας τα πολιτικά θεσμικά ωφέλη που έχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ για την ε, ομιλία σας και για την στράτευσή σας. Θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα τον αρμόδιο επίτροπο, κύριο Χωακίμ Αλμούνια. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Δέκα χρόνια μετά την έναρξή του είμαι βέβαιος ότι συμφωνώ με τη μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και μπορώ να πω ότι ως Ευρωπαίος είμαι υπερήφανος για την επιτυχία του ευρώ. Και θέλω να συγχαρώ το Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία αυτή που ανέλαβε σήμερα εδώ ε, στην αίθουσα ε, της ε, Ολομελίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εορτάσουμε τη δεκάτη επέτειο του κοινού μας νομίσματος. Το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και η Οικονομική Ένωση είναι σίγουρα μεγάλη επιτυχία, αναφυσβήτητη. Τα τελευταία δέκα χρόνια το ευρώ έφερε πολλά ευεργετήματα ε, σε όλα τα μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωζώνη και εξακολουθεί να το πράττει σήμερα ε, μεσού τη βαθιά ε, χρηματοπιστωτική κρίση. Είναι σύντομο το διάστημα τη δεκαετία, αλλά απέκτησε άξια φήμη το ευρώ για σταθερότητα και ισχύ. Είναι το δεύτερο παγκόσμιο νόμισμα χάρη στο ρόλο που διαδραματίζει στη διεθνή οικονομία και χάρη σε αυτό ήδη συγκρίνεται με το δολάριο σε ορισμένες πτυχές ως εργαλείο διεθνούς εμπορίου και μέσων πληρωμών στα διεθνή χρηματοπιστωτικά. Κυρίως όμως το ευρώ αποτελεί τμήμα της καθημερινότητας 330 περίπου εκατομμύριων πολιτών σε 16 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι έχουμε στα πορτοφόλια μας το σύμβολο αυτό της κοινή ευρωπαϊκής ταυτότητας. Διότι το ευρώ εκτός από νόμισμα είναι και κομβικό στοιχείο του ευρωπαϊκού εγχειρήματο και σχεδίου που συγκεκριμένα μας θυμίζει τα ωφέλη που έχουμε από τη διαδικασία ολοκλήρωσης που ε, ξεκίνησε εδώ και 50 και πλέον έτη το ευρώ μας εξασφαλίζει χαμηλό πληθωρισμό, χαμηλά επιτόκια με ένα μακροοικονομικό πλαίσιο που προσανατολίζεται στη σταθερότητα. Το ευρώ μας δίνει σαφή όθηση στο εμπόριο και στις επενδύσεις μεταξύ των κρατών μελών. Το ευρώ <coughs> επέτρεψε τη δημιουργία 16 εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης τα τελευταία 10 χρόνια στην Ευρωπαϊκή ε, ε, Ήπειρο και τριπλάσιο από την προηγούμενη δεκαετία. Υποστήριξε και ανάπτυξε την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, προστάτευσε την Ευρώπη από τους εξωτερικούς ε, τριγμούς και ήταν σύμβολο όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Σίγουρα η κρίση είναι δοκιμασία για το ευρώ, αλλά πλανώνται εκτρά εκεί που νομίζουν ότι η ΟΝΕ δεν είναι προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Το αντίθετο. Εάν δεν είχαμε νόμισμα, οι αντικσοότητες και οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης θα ήταν πολύ περισσότερες. Πολλά κράτη-μέλη σήμερα θα ε, είχαν μεγάλη πτητικότητα στις ισοτιμίες των νομισμάτων και μπορεί να ήταν και θύματα κερδοσκοπικών επιθέσεων κατά των νομισμάτων τους. θα είχαν ε, πολύ μεγαλύτερα ελλείμματα και ε, δημόσια και χρέη και θα είχαν λιγότερες δυνατότητες αντιμετώπισης ε, της κρίσης αυτής. Από το 2005 η αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητα βοήθησε τα κράτη-μέλη να εξηγιάνουν τα δημόσια οικονομικά του και το 2007 είχαμε τα πιο ε, χαμηλά δημόσια ελλείμματα τη τελευταία 20 πενταετία. Και μπορούμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε με καλύτερου όρου την κρίση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδειξε μια στάση και συμπεριφορά που ενίσχυσε και μόνο τη ε, ισχυρή και στέρεη φήμη που είχε ήδη από την αρχή το ευρώ. με αποφασιστικότητα έλαβε τα απαραίτητα μέτρα και ηγήθηκε στη συνεργασία των υπολείπων κεντρικών τραπεζών των βιομηχανικών κρατών και η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα μας ε, καθοδήγησε το τελευταίο διάστημα και συνεισέφερε ουσιαστικά για να απευθυνθεί μια τεράστια χρηματοπιστωτική κατάρρευση. Η οικονομική κατάσταση δεν είναι εκείνη που θα επιθυμούσαμε για να εορτάσουμε την επέτειο αυτή σήμερα. Αλλά τα γεγονότα και εξελίξεις τονίζουν ακόμα περισσότερο και όσο ποτέ τα ε, ευεργετήματα και τα πλεονεκτήματα της Ευρωζώνης. Είναι όλο και πιο ελκυστική αυτή η ζώνη για νέες χώρες. Το ζήσαμε στην Πρατισλάβα την περασμένη εβδομάδα, όταν καλωσορίσαμε τη Σλοβακία στους κόλπους της Ευρωζώνης. Είναι το 16ο μέλος της οικογένειας του Ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τα κράτη-μέλη στην Ευρωζώνη, την Ευρωομάδα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ε, σε συνεργασία πάντα με τη διεθνή κοινότητα να ξαναφέρουμε τις οικονομίες μας στο μονοπάτι της αηφόρου ανάπτυξης και της ε, ευημερίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση που παρουσίασε πριν από μερικούς μήνες για την πρώτη δεκαετία του ευρώ κάνει προτάσεις και αυτή η έκθεση άλλωστε συζητήθηκε πρόσφατα στο κοινοβούλιο σας και αυτά τα συμπεράσματα ισχύουν πολύ περισσότερο σήμερα από ό,τι την περασμένη άνοιξη. Δημοσιονομική επαγρύπνηση, ε, μακροοικονομικά στοιχεία, συνεργασία ε, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με τη μακροοικονομική πολιτική, εξωτερική προβολή του ευρώ και βελτίωση της διαχείρισης στην ΟΝΕ είναι και παραμένουν οι άξονες στους οποίους στηρίζεται η δεύτερη δεκαετία του ευρώ ε, ελπίζουμε να έχει τουλάχιστον ε, αντίστοιχες εξίσου πολλές επιτυχίες με την πρώτη. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας θα ήθελα να ποτίσω ένα φόρο τιμής στο όραμα και στη φιλοδοξία των ιδρυτών, των πατέρων του ευρώ που με τη φαντασία τους και τη δράση τους, την αποφασιστική, μας άφησαν, μας κληροδότησαν ένα νόμισμα για το οποίο όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούμε να αισθανόμαστε περήφανοι. Τώρα θα πρέπει να διαφυλάξουμε τα θεμέλια αυτή τη επιτυχία. Η κρίση άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για την παγκόσμια οικονομία, όπου η Οικονομική και Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο υπέρ των συμφερόντων και των ε, φιλοδοξιών που ενώνουν όλου του Ευρωπαίου. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την ομιλία σας και για την προσπάθεια που καταβάλλετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιτυχία των θεμάτων αυτών. Τώρα, με μεγάλη μας χαρά, θα ήθελα να ακούσουμε τον πρώην πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και πρώην συνάδελφό μας, κύριο Βαλερίζη Καδεστά. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριοι Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Όσοι εργάστηκαν για την γέννηση του Ευρωπαϊκού Νομίσματος, σας είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες κύριε Πρόεδρε Hans Gert Pöttering και σε εσά, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές για την καλή πρωτοβουλία που αναλάβατε να γιορτάστε την δεκάτη επέτειο της γέννησης του ευρώ. Είμαι μεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι είναι καλύτερα να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός ε, των τελετών και των εορτασμών, αλλά αυτή είναι δικαιολογημένη διότι είναι η μεγαλύτερη συμβολή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ενοποίηση από την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψήφο το 1979. Ο δρόμος υπήρξε μακρύς και επίπονος και ίσως αυτή η συγκέντρωση, η χαρούμενη και η εγκάρδια δεν αντανακλά πλήρως την σημασία του δρόμου αυτού. Θα ήθελα να ποτίσω φόρο τιμή σε αυτούς που χάραξαν αυτό το δρόμο και τον ακολούθησαν. Μπορούμε να βρούμε ε, την μακρινή προέλευσή του στην έκθεση του, προ, του Πιερ Βερνέρ, του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, του Προκατόχου σας το 1970 αλλά είναι η νομισματική κρίση των επομένων ετών ε, και η ε, μεταβλητότητα των ισοτιμιών των νομισμών που ε, ενέτειναν την κίνηση αυτή. Ενώ ήταν σταθερές οι ισοτιμίες δεν υπήρξαν διαταραχές στην κοινή αγορά. Από την στιγμή όπου ήταν μεταβλητές οι ισοτιμίες τέθηκε το πρόβλημα μετά τις ατυχείς προσπάθειες δημιουργίας ενός νομισματικού ε, φυσιδιού είναι η όθηση η γερμανο της, ε, του 1975 και της δεκαετίας του 80 που οδήγησαν στην Βρέμη, σε αυτήν την βόρεια πόλη της Γερμανίας, την απόφαση δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος και της εισαγωγής του Εκιού, που ήταν το πρόδρομος ε, του ε, ευρώ. Αυτή η προσπάθεια συνοδεύθηκε και στηρίχθηκε από τους εταίρους μας του Μπενελούξ και της Ιταλίας μετά από ε, μια περίοδο ε, ύπνωσης μεταξύ του 85 και του 88 ο δρόμος προς τα μπρος συνεχίστηκε με την δημιουργία από το Συμβούλιο της Επιτροπής με επικεφαλής τον Ζακ Ντολόρ που κατέληξε στην υπογραφή της συνθήκης του Μάστριχτ και θα θέλα να χαιρετήσω τους ε, σκαπανείς, τους πρωτοπόρους που εργάστηκαν στο δρόμο αυτό, στην διάρκεια αυτή, στη διαδρομή αυτή, τον καγκελάριο Χέλμουτ Σμιτ και τον Λαμφστάιν, τον υφυπουργό, τον ε, κυβερνήτη, ε, το διοικητή της Τράπεζας Γαλλίας Ραπιέ που ήταν μαζί με τον Ρόμπερ Σουμάν συντάκτης της διακήρυξης, τον κύριο Λαμφαλούση, ο οποίος προσέφερε τη τις γνώσεις του, τις μοναδικές του γνώσεις στις εργασίες της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση που δημιουργήσαμε με τον Χάιλμουτ Σμιτ για να αναθερμάνουμε ε, την όλη αυτή η προσπάθεια. Ο πρόεδρος Ζακ Ντολόρ, ο οποίος ανέλαβε τη σκητάλη και τέλος ε, τους διαπραγματευτές και αυτούς που υπέγραψαν τη συνθήκη του Μάστριστ που συνέταξαν ένα πάρα πολύ καλό κείμενο το οποίο υπάρχει από τότε και πρέπει να τονίσουμε την αποφασιστικότητα του καγκελαρίου Helmut Kohl και του ε, Προέδρου Φρανσουά Mitterrand, όπως επίσης και των συναδέλφων τους. Σε όλους αυτούς, σήμερα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε αυτήν τη δεκάτη επέτειο που γιορτάζεται σε εποχή κρίσης, τι μπορούμε να πούμε για το ευρώ. Ε, σε τι μπορούμε να πιούμε κατά κάποιο τρόπο. Πρώτα απ' όλα η επιτυχία του ευρώ ξεπέρασε τις προσδοκίες όχι μόνο όλων των αντιπάλων του ευρώ αλλά ακόμα και των υπερμάχων του ευρώ. Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες, διότι μου δώσατε μόνο πέντε λεπτά ε, και οι μεγάλες συζητήσεις που είχα ε, στην, ε, το 1995 και μέχρι το 2000, οι συζητήσεις που είχα με τους ειδήμονες μου έδειξαν ότι όλοι εξέφραζαν μεγάλες αμφιβολίες για το ευρώ και την επιτυχία του. Σε 10 χρόνια το ευρώ έγινε το δεύτερο παγκόσμιο νόμισμα, διεθνές νόμισμα και ένα από τα νομίσματα που την χάνει μεγάλου σεβασμού. Η καλή διαχείριση του ευρώ το κατέστη ασπίδα κατά της κρίσης και βάση ε, για μια ανάπτυξη χωρίς πληθωρισμό. Χωρίς την ύπαρξη του ευρώ, η υπηρετική Ευρώπη σήμερα θα κλειδονιζόταν ε, με έναν ανεμοστρόβιλο νομισματικό ε, που θα ερχόταν να επιδεινώσει την οικονομική κρίση. Περιμένουμε από την νομισματική πολιτική να προσπαθήσει να συγκρατήσει μέσα στα όρια των δυνάμεων του νομίσματος ε, τις καταθλιπτικές συνέπειες της κρίσης και να προετοιμάσει την επάνωδο. Δεν έχουμε ακόμα ετοιμαστεί για την επάνωδο, μια επάνωδο στην ανάπτυξη, στην οικονομική μεγέθυνση χωρίς πληθωρισμό όταν ε, θα τελειώσουμε με, τις, με τα μεγάλα δημόσια ελλείμματα και την υπερχρέωση στην οποία οδήγησε η κρίση και σας εμπιστευόμαστε τους ηγέτες, το ηγετικά στελέχη και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι θα βρουν το δρόμο να τα επιτύχουν αυτά, διότι κατά τη διάρκεια της κρίσης επέδειξαν την πραγματογνωμοσύνη τους και σεβόμαστε την αποφασιστικότητά τους και την ανεξαρτησία τους. Δύο παρατηρήσεις για να κλείσω. Ας προσέξουμε όμως διότι δεν πρέπει να δώσουμε στο ευρώ μια παγκόσμια διάσταση που θα κολάκευε τη ματαιοδοξία μας βεβαίως και που θα πολλαπλασίαζε τους κινδύνους μας. Το ευρώ είναι το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Υπήρου και για να εκφράσουμε την ιδιαίτερη κουλτούρα του ε, τους, γιατί που είναι ο λόγος της ε, σταθερότητάς του μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας των άλλων νομισμάτων. Δεν νομίζω όμως ότι θα πρέπει να, να περιμένει πολύ η κοινή γνώμη για ε, την ρύθμιση της οικονομικής ζώνης του ευρώ. Μου φαίνεται ότι εδώ θα μπορούσαμε Σύμφωνα με το άρθρο 106, παράγραφο 5 της συνθήκης του Μάστριχ, θα μπορούσαμε εδώ να καταφύγουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να μπορέσει να, να, ε, να οδηγήσει, να διευθύνει αυτήν ε, την ε, ρύθμιση διότι χρειαζόμαστε αυτές τις γνώσεις, χρειαζόμαστε ένα χρονοδιάγραμμα αποφάσεων που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε ε, να προσδιορίσει. Εσείς ε, ο, και, ο, και που ο κύριος Γιούγκερ θα μπορούσε μετά ε, να επικυρώσει. Θα κλείσω κύριε Πρόεδρε λέγοντας ότι το σύμβολο της ενοποίησης, της ολοκλήρωσης που είναι η επιτυχία του ευρώ πρέπει να μας δώσει το θάρρος να προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτή την οικοδόμηση στην οικοδόμηση αυτής της Ευρώπης, η οποία είναι όλο και περισσότερο ενωμένη, που μας προτείνουν οι συνθήκες και που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και να διαμορφώσουμε στην ητοπάθεια της αποτυχίας ας αντιτάξουμε την δυναμική της επιτυχίας και η επιτυχία εδώ σήμερα έχει μια ωραία λέξη, ονομάζεται ευρώ. Ευχαριστώ πολύ σε όλες τις γλώσσες. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Κύριε Πρόεδρε, στα γαλλικά ο του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε όχι μόνο για την ομιλία σας, αλλά και όλους ιδιαιτέρως για την προσωπική σας ιστορική συνεισφορά. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε Ζησκάρδιστα. Äh, Ακολουθούν οι δύο εισηγητέ, πρώτα η πρόεδρο τη Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, κυρία Περβά ε, Μπερέ, και στη συνέχεια ο Βέρνερ Λάγκερ. Παρακαλώ, κύριε Μπερέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ευρώ είναι επιτυχία ενός οράματος, μιας πολιτικής βούλησης. Δεν είναι καρπός της αγοράς. Είναι η απόδειξη εκείνων που μπορεί καλύτερα και ξέρει καλύτερα να δημιουργεί η Ευρώπη όταν κινητοποιούνται όλοι. Θα ήθελα βεβαίω εδώ να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω εξ ονόματός μας, εξ των παιδιών μας και όλων μας τους ιδρυτές πατέρες και τους εμπνευστές αυτής της επιτυχίας. Τον Πιεβερνέ που βρίσκεται τον καγκελάρη Χελμουντ τον πρόεδρο Ζισκάρτεστεν, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Λόρ, ε, τον κύριο Κόλ, τον κύριο Μίτεραν, ε, τον Λαμφαλουσί, τον Μασκόπα, Φιλίπ Μεστάτ και όλους εκείνους που ε, ξεχνώ. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω τη δράση των προκατόχων σας κύριε Πρόεδρε και των δικών μου. Ο Κάλφον Βόγκαου είναι ακόμα ε, συνάδελφος και η Κρίστα Ράντζιο Πλάτ παρευρίσκεται επίσης. Γιατί η δράση του Κοινοβουλίου αυτού ήταν αποφασιστική. Τη στιγμή της μετάβασης στο ευρώ έπρεπε να ασχοληθούμε όχι μόνο με τη μεταφορά των λογιστικών στοιχείων στις τράπεζες αλλά και με τους πολίτες τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ε, συνηθίσουν στο ευρώ, να υιοθετήσουν το ευρώ, να το αγκαλιάσουν αυτό το νέο νόμισμα, ε, νόμισμά τους. Και νομίζω θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και να χαιρετήσουμε και το ρόλο του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να εκφράσω και την ικανοποίησή μου που η ε, επέτειος αυτή εορτάζεται εδώ πανηγυρικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον οίκο της Δημοκρατίας, στον οίκο των Ευρωπαίων πολιτών. Διότι το ευρώ είναι πρώτα απ' όλα υπόθεση όλων και μετά υπόθεση των τραπεζών. Είναι υπόθεση των Ευρωπαίων και μας το λέγουν. Ορισμένες κυβερνήσεις δεν θέλουν η Ευρώπη να έχει σύμβολα. Οι Ευρωπαίοι όμως οι ίδιοι υιοθέτησαν το ευρώ ως σύμβολο ε, ε, του ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως δεν έχουμε όλοι ευρώ. Στην αρχή είμαστε 11, τώρα είμαστε 16. Περιμένουν να έρθουν και άλλοι στην οικογένεια του ευρώ. Ωστόσο έχω την εντύπωση ότι η κρίση αυτή καλεί ορισμένους να αναθεωρήσουν τι τάσει τους και τη συμμετοχή τους ή όχι στην Ευρωζώνη. Ποια καλύτερη απόδειξη επιτυχίας. Η Ευρώπη συχνά προχωράει όταν δοκιμάζεται η αποτελεσματικότητά της. Και επί τη ευκαιρία της επαιτίου της δεκάτης του ευρώ βλέπουμε ότι έχει θετικό απολογισμό. Ορισμένοι που ήταν κάπως επιφυλακτικοί και διστακτικοί σήμερα θα μπορούσαν να κρούσουν τι θύρε ε, της Ευρωζώνης. Και δεν μπορούμε παρά να τους ενθαρρύνουμε να το πράξουν υπό τους όρους που ορίζει η συνθήκη που ποτέ δεν αναθεωρήθηκαν και είναι χρήσιμοι όροι για να μπορέσει η Ευρώπη στο νομισματικό και οικονομικό τομέα να προοδεύει στους δύο αυτούς πυλώνες και στην ευάθυνση και στη διεύρυνση. Αλλά μια επέτειος είναι και ε, μια στιγμή που μας επιτρέπει να κοιτάξουμε προς το μέλλον. Το ευρώ με τον πλούτο και την εμπειρία των 10 ετών θα πρέπει σήμερα να ξεκινήσει νέε προσπάθειες. Όχι ότι δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με αυτές, αλλά ε, ε, γιατί ακόμα εκκρεμούν διάφορα θέματα. Στην οικονομική συνεργασία ο Ζων Κλοντ Ιούνκερ περιέγραψε την έλλειψη ευρωπίας που ζούμε σήμερα. Δεν είναι φυσιολογική αυτή. Και σήμερα στην κρίση γνωρίζουμε όλοι ότι αν είχαμε προοδεύσει στην Οικονομική Ένωση όσο προεδρεύσαμε στην Νομισματική Ένωση, τότε σήμερα θα είμαστε ακόμα καλύτερα εφοδιασμένοι. Α βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και τα διδάγματα. Δεν μπορούμε να, να βλέπουμε μόνο την ποσότητα των ελλημάτων και όχι την ποιότητα των οικονομικών πολιτικών. Θα πρέπει οι κυβερνήσει να συνεργάζονται. Δεν είναι φυσιολογικό τα κράτη-μέλη να δανείζονται με τόσο διαφορετικά επιτόκια ενώ έχουν ε, το ίδιο νόμισμα και το ίδιο επιτόκιο από την Κεντρική Τράπεζα. Το ίδιο ισχύει και για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών, Αναφέρθηκε στο άρθρο 105 εδάφιον 6 ο πρόεδρος της Είναι η κοινή μας βάση και σε αυτή θα προχωρήσουμε όλοι. Ένα από τα εντάγματα της κρίσης είναι να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να διαδραματίσει ένα ρόλο στην εποπτεία. Δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε την εποπτεία των χρηματαγορών από την ε, εποπτεία της μακροοικονομίας και τη συνετή διαχείριση. Θα πρέπει όμως και εμείς οι πολιτικοί να σκεφτόμαστε την ισορροπία. Μπορεί ε, αν ενισχυθεί η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να δούμε και τη διαφορετική θεσμική ισορροπία και πώς θα διαμορφωθεί αυτή στο μέλλον. Τελευταία παρατηρήση για το διεθνή ρόλο του ευρώ. Συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να διεκδικούμε το εξωφρενικό ε, προνόμιο να είμαστε ένα νόμισμα αποθεματικού. Μα δέκα χρόνια κάναμε για να ε, ε, φτιάξουμε το ευρώ. Δέκα χρόνια μετά το ευρώ δεν μπορούμε να χωλένουμε διεθνώς ε, στη διεθνή χρηματοπιστωτική πραγματικότητα και να μην είναι καλύτερο οργανωμένο το σύστημα. Το ευρώ τέλος είναι πολύ περισσότερο από ένα νόμισμα. Γι' αυτό είναι μίζον αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ένα εργαλείο στην υπηρεσία των πολιτών που ζουν την πιο σοβαρή κρίση των τελευταίων ετών και, ετών. και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ε, αυτό το καταπληκτικό επίτευγμα και σύμβολο ώστε οι πολίτες να περάσουν την κρίση αυτή με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάγκεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δέκα χρόνια ευρώ. Πραγματικά αυτό αποτελεί λόγο για να εορτάσουμε. Όποιος θα μας έλεγε πριν από δέκα χρόνια ότι θα είχε τέτοια επιτυχή πορεία το ευρώ Νομίζω ότι ε, πολλοί θα τον περιγελούσαν. Πολλοί εργάστηκαν για ε, την επιτυχία αυτή. Θυμούμε πολλούς βέβαια που ήταν επιφυλακτικοί, που μιλούσαν για θνησιγενή εγχειρήματα κλπ. Σήμερα γνωρίζουμε ότι υπήρξε ένα όραμα το οποίο είχε πολλούς πατέρες, θύμισαν οι προηγούμενοι που ε, μίλησαν ποιοι ήταν όλοι αυτοί. Μιλώ και για ένα πρώτο μια πρώτη προσπάθεια που ήταν η Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα, την έκθεση Delors για την Νομισματική Ένωση σε τρία στάδια, την συνθήκη του Μάστριχτ, μόνο δύο χρόνια μετά από την πτώση του τείχους. Πολλοί συνεργάστηκαν ώστε σήμερα το ευρώ να είναι επιτυχία. Κυρίε και κύριοι, νομίζω ότι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η κυρία Μπερέ το είπε ως πρόεδρος της Επιτροπής Νομισματικών στην παρούσα περίοδο και από το 1994 όταν άρχισε να εφαρμόζεται η συνθήκη του Μάστριχτ και μέχρι το 2002, μέχρι δηλαδή την εισαγωγή των νομισμάτων, των κερμάτων και των χαρτονομισμάτων, με πολλές ε, εκθέσεις και ε, προτάσεις και ψηφίσματα συνέβαλε στην προσπάθεια αυτή και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους δύο τότε Προέδρους της Επιτροπής Νομισματικών, Κάλφον Βόγκαου και Κρίστα Ράντζιο Πλάτ, ε, που εξεπροσώπησαν το Κοινοβούλιο και προς τα έξω και προσέφεραν την απαραίτητη κοινοβουλευτική υποστήριξη στις προσπάθειες των τότε κυβερνήσεων. Σήμερα, υπό την Προεδρία της ε, κυρίας Μπερές, συνεχίζει η Επιτροπή Νομισματικών την ίδια προσπάθεια και εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου προς τα έξω. Γνωρίζετε ότι στις 18 Νοεμβρίου υιοθετήσαμε έκθεση όπου αναφερόμαστε και στις επιτυχίες αλλά και στις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το ευρώ σε συμπλήρωση των όσων είπε η κυρία Μπερέ, θα προσφέρω και εγώ ορισμένε σκέψει. Το ευρώ είναι μεγάλη επιτυχία και είναι και μοναδικό εγχείρημα. Μια κεντρική πολιτική χρήματο υπό την κατεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μια αποκεντρωμένη δημοσιονομική πολιτική. Είναι σημαντικό η διασύνδεση μεταξύ των δύο αυτών επιπέδων ευθύνη στο μέλλον και η διασύνδεση αυτή είναι το σύμφωνο σταθερότητα να διατηρηθεί και στο μέλλον. Γιατί χωρί σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη, χωρί καλύτερο συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών θα, αντιμετωπίσει το ευρώ και στο μέλλον βαρύτατου κινδύνου. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση ιδίω προς τις ε, χώρε μέλη τη Ευρωζώνης αλλά και σε όλε τι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να διατηρήσουν αυτή την πειθαρχία, να διατηρήσουν αυτή τη συντονισμένη συνεργασία και να την πάρουν περισσότερο σοβαρά υπόψη τους από ότι κάποιες περιπτώσεις στο παρελθόν. Το ευρώ συμπίεσε τον πληθωρισμό και μάλιστα σημαντικά, δίνοντας έτσι εμπιστοσύνη στον κόσμο. Και έγινε και το δεύτερο νόμισμα αποταμίευσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει ενισχύσει τις δομές στις χώρες μέλη και προσφέρει και την δυνατότητα να ισχυροποιηθούν οι επιχειρήσεις και τα κράτη μέσα σε μια περίοδο κρίσεων τα θεσμικά όργανα της Ευρωζώνης, το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ, η Ομάδα Ευρώ, αλλά και άλλοι θεσμοί έχουν δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις επειδή λειτουργήσαν, επειδή υπήρχαν και επειδή λειτουργούσαν. Και επειδή λειτουργούσαν ανεξάρτητα, αλλά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε να μπορούν και σε συνθήκες κρίσεως να αντιδρούν με ταχύτητα. Έχουμε το ευρώ και ως μοχλό για την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής ενιαίας Αγοράς. Και νομίζω ότι τα πολιτικά διδάγματα από την κοινή αυτή επιτυχία είναι ότι χώρες με ισχυρό νόμισμα και μια ισχυρή ενιαία αγορά έχουν φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο ενοποίησης το οποίο εξασφαλίζει την ειρήνη και την ευημερία. Όμως το ευρώ δεν θα είναι αυτονόητο και για το μέλλον. Υπάρχει ένα πλήθος απαιτήσεων για το μέλλον πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Ε, η σύγκληση των διαφόρων οικονομιών, για παράδειγμα, για την εξέλιξη των μισθών, για τα ελλείμματα, εκεί υπάρχουν και κίνδυνοι που δεν πρέπει να αποσιωπηθούν, έστω και μέσα στην εορταστική σημερινή ατμόσφαιρα. Και ένα άλλο θέμα, ότι οι διαφορετικές εξελίξεις των επιτοκίων για τα κρατικά δάνεια βλέπουμε ότι αυξάνει πάλι, ανοίγει πάλι η ψαλίδα. Αυτά ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα προβλήματα στις ε, χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Και σε ό,τι αφορά την επέκταση της ε, ζώνης ευρώ δεν πρέπει να υπάρξουν εκεί εκπτώσεις, καμία έκπτωση. Οι χώρες οι οποίες θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωζώνης πρέπει να εκπληρούν όλα τα κριτήρια της συνθήκης του Μάστριχτ. Κυρίε και κύριοι, νομίζω ότι το ευρώ έχει γίνει αποδεκτό από τους πολίτες, χέρι της παγκόσμιας εμπιστοσύνης, έχει περάσει τις ε, πρώτες δοκιμασίες και αποτελεί όντως μια μοναδική συνεισφορά στην διαρκή ενοποίηση των προσπαθειών των λαών των, της Υπήρου μας. Και γι' αυτό μπορούμε να είμαστε νομίζω υπερήφανοι όλοι. Σας ευχαριστώ κύριε Λάγκεν. Ακολουθούν οι πολιτικές ομάδες. Πρώτα ο κύριος Σον Κλοντ Ποζέ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Γκοζέ, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολλά πράγματα ελέγχθησαν και ήταν σωστά μέχρι τώρα. Η, μέσα σε 10 χρόνια το ευρώ έγινε το, σύμβολο, το ισχυρό σύμβολο της Ευρώπης. Και όμως ο, το γεγονός ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κοινό νόμισμα ε, τα θεμέλια του οποίου είχαν ε, ξεκινήσει το 1968 στη συνθήκη της Βρέμης και τη δημιουργία του ΕΚΙΟΥ ε, αυτό ήταν μια μεγάλη φιλοδοξία και όσοι συμμετείχαν στην απόφαση αυτή θα πρέπει να τους συγχαρούμε θέρμα και να τους ευχαριστήσουμε. Η δημιουργία του ευρώ είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η Ευρώπη είναι ικανή, ε, εάν και εφόσον υπάρχει ισχυρή πολιτική θέληση, να υιοθετήσει μακροπρόθεσμες αποφάσεις ε, για ένα ε, μέλλον μεγάλων προσδοκιών και πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα πάρα πολύ θετικό στη συγκυρία την οποία ζούμε. για τους πολίτες μας μέχρι πρόσφατα το ευρώ ήταν λίγο αντιφατικό. Για όσους ε, ταξιδεύουν ε, το, το προτέρημα ενός ενιαίου νομίσματος ήταν προφανές. Όμως ε, για τους υπόλοιπους το ευρώ μεταφράστηκε σε υψηλές τιμές. Όμως είδαμε ότι ο, ενώ τα επίσημα στοιχεία έδειχναν ότι χάρη στην δράση της Κεντρικής Τράπεζας νομισματική σταθερότητα υπήρχε, υπήρξε ένας ε, προφανής πληθωρισμός των τιμών. Ε, γιατί ορισμένοι στρογγύλεψαν τις τιμές σε ευρώ, σε κάποια προϊόντα και οι καταναλωτές δεν ήταν αρκετά ε, προσεκτικοί. Επίσης ακούσαμε τα σχόλια κάποιων βιομηχανιών που παράγουν στην ε, Ευρώπη και εξάγουν και εκεί είχαμε ε, διάφορες δυσκολίες όταν ε, λόγω της ισοτιμίας με το δολάρια. Και προφανώς η ισοτιμία ήταν πάρα πολύ ψηλή. Σήμερα όμως η κρίση τροποποίησε όλες αυτές τις εκτιμήσεις. Όλοι θεωρούν ότι το ευρώ είναι ένα αποφασιστικό στοιχείο έτσι ώστε να περιορίσουμε τις ευρωπαϊκές συνέπειες μιας κρίσης την οποία ζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης ήταν η πιο δραστήρια. Οι αποφάσει ε, τη οι πάρα πολλέ ε, σωστέ χαιρετίστηκαν ε, από όλου. Ποια θα ήταν η κατάσταση εάν τα διάφορα κράτη έπρεπε να υπερασπιστούν από το καθένα το δικό του νόμισμα. Οι υποτιμήσει θα ήταν αναπόφευκτε. Δεν θα αποφεύγαμε μια νομισματική κρίση. Το ευτυχέ αποτέλεσμα του ευρώ θα πρέπει να μα οδηγήσει να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και να σεβαστούμε τι αρχέ του Συμφώνου σταθερότητα και ανάπτυξη. Βέβαια, βέβαια στην ε, περίοδο την οποία να ζούμε θα μπορούσαμε να ε, δεχτούμε και θα πρέπει να δεχτούμε κάποιες εξαιρέσεις. Όμως οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να είναι προσωρινές και θα πρέπει να έχουμε σαν στόχο τα ισορροπημένη οικονομική, τα οικονομία των κρατών. Η ισορροπία αυτή θα πρέπει να ε, τονίσει και να προβάλλει, την, να προβάλλεται στο μέλλον. Θα πρέπει να προχωρήσει η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη. Αυτές, αυτά τα δύο στηρίζονται και στην σταθερότητα του ευρώ του νομίσματός μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκοζές, ακολουθεί ο Ρομπέρ Γκέμπελς από τους Σοσιαλδημοκράτες για πέντε λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτούς τους καιρούς αφεβαιότητας είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να υπολογίζει σε μια σταθερή αξία, το ευρώ. Στην προπαρασκευαστική φάση είχα την ευκαιρία να προετοιμάσω ε, το ευρώ σε ένα σκαμνάκι στο ΕΚΟΦΗΝ και μπορώ να σας πω ότι είχαν μεγάλες επιφυλάξεις ε, τα κράτη-μέλη. Αλλά τελικά συμφώνησαν στην Ευρωζώνη, στην Ευρωομάδα και προχώρησαν σε μια ενισχυμένη συνεργασία που είναι ακόμα αυτή ε, θεσμοθετηθεί. Ορισμένες χώρες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε απτά χειροπιαστά αποτελέσματα. Μιλώ για το Σέγγεν και τη συνθήκη που ξεκίνησε από πέντε χώρες, τη Γαλλία του Μιτερά, τη Γερμανία του Κόλ και τις χώρες Μπενελούξ. Σήμερα έχει μπει στο Σέγγεν μέχρι και η Ελβετία, αλλά οι Ιρλανδοί και οι Βρετανοί ε, ακόμα διστροπούν προς την Ευρώπη των πολιτών και δεν συμμετέχουν. Ο Μιτεράν και ο Κόλ ήταν επίσης οι πολιτικοί γονείς της Ευρώπης. Ε, βέβαια η νομισματική ένωση έχει πολλούς πατέρες τη αρχή γενομένη από τον Ζακ Ντελό. Το πρώτο δίδαγμα που θα ήθελα να εξάγω είναι ότι όλοι εκείνοι που θέλουν μια καλύτερη Ευρώπη δεν θα πρέπει να φοβούνται τη διακυβερνητική συνεργασία και δράση. Ιδιαίτερα όταν ε, έχουμε... Ε, συμμαχία κάποιων κρατών που θέλουν πραγματικά να προωθήσουν την Ευρώπη. Η συνθήκη του ΠΡΟΥΜ που επιτρέπει την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος είναι ε, άλλο ένα εύγλωτο παράδειγμα της ενισχυμένης αυτής θετικής συνεργασίας για την Ευρώπη. Τη στιγμή που η συνταγματική συνθήκη έχει ενταφιαστεί μετά από το όχι ε, μια περίεργη συμμαχία Γάλλων και Ιρλανδών και η μήνυ συνθήκη τη που ε, ε, στην Ιρλανδία και στην Τσεχική Δημοκρατία γνωρίζει δυσκολίες και ε, δυστοκίες, θα πρέπει να δούμε πώς θα ενισχυθεί η ενισχυμένη συνεργασία. Η ε, ελκυστικότητα πάντως του ευρώ διατηρείται στο ακέραιο. Μετά τη Σλοβενία ήρθε και η Σλοβακία. Άλλοι ανησυχούν και δεν θέλουν να ε, μπορέσουν να υποφεληθούν από τα ωφέλη του ε, ευρώ. Ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε γιατί να μην μπορούμε και εμείς να εκμεταλλευτούμε το ευρώ ενώ η λίρα έχει αρχίσει να καταραίει. Και, ε, μετά τον Ντόισπερκ, τον Τρισέ, τον Τρισέ και άλλους έχουμε περάσει σε δεύτερο επίπεδο αποθεματικών ανά τον κόσμο σε ευρώ. Βέβαια παραμένει βασιλιάς και κυρίαρχος το δολάριο και παραμένει η αξία καταφύγιο για τις οικονομίες, αλλά όταν οι ΗΠΑ αποφάσισαν να χρηματοδοτούν το ακριβό τον ακριβό τρόπο ζωή τους ε, ει βάρο ολόκληρου του κόσμου υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βλέπουν ότι το δολάριο δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις υποσχέσεις και τι δεσμεύσει τους. Τώρα ίσως κάποιοι φοβούνται ότι περνούμε σε ένα διοπόλιο πλέον δολαρίου και ευρώ. Με προσαρμογή βέβαια των ισοτιμιών όταν όμω έχουμε ε, ύφεση γενικευμένη χρειάζεται σταθερότητα, ασφάλεια στον κόσμο, βεβαιότητες. Το ευρώ θα αποτελέσει ένα κεντρικό στοιχείο αυτής της νέας σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε ό,τι μπορούσε απέναντι στην διεθνή δημοσιονομική κρίση, ε, χρηματοοικονομική κρίση που ήταν made in USA. Όπως είπε ο Σακτουλόχ, ήταν η ασπίδα ολόκληρου του κόσμου το ευρώ. Η Ευρώπη μέχρι τώρα δεν έχει μπορέσει να δώσει αρκετό δυναμικό, αρκετή δύναμη στην ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική. Μόνο η νομισματική αντιμετωπίζει ε, με την ε, λειτουργία του ευρώ. Πλην όμως οι πραγματικοί οικονομικοί φορεί παραμένουν τα κράτη-μέλη και μάλιστα δρούν κατακαιρματισμένα. Η οικονομική, οικονομική δύναμη όμως των 27 κρατών ε, μαζί θα μπορούσε να εξασφαλίσει θαυματουργές λύσεις και αποτελέσματα. Ε, η λέσχη όμως του ευρώ του Ζων Κλοντ Γιουνκέρ παραμένει μόνο μία και κλεισμένο των θυρών λέσχη συνομιλιών ε, για θέματα οικονομικά. Εγώ ήμουν παρόν ε, σε κάποιες προσπάθειες των Υπουργών Λαφοντέν, Στροσκάν και άλλων ε, που προσπαθούσαν να βρουν λύσεις οικονομικές ε, με το ευρώ μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ο Βιμ Ντοϊσπερκ έδωσε τη σκληρή απάντηση ποτέ δεν θα υπάρξει εξάντε συντονισμός με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάντοτε εξπόστρα θα αντιδράτε εκ των υστέρων στις αποφάσεις των ε, κυβερνήσεων. Όντως, όντως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι και παραμένει ανεξάρτητη στην ε, διαξαγωγή της νομισματικής της πολιτικής. Αυτή η ανεξαρτησία όμως δεν απαγορεύει τον επικοδομητικό διάλογο μεταξύ θεσμικών οργάνων. Δεν απαγορεύει να προστατεύουμε όλοι από κοινού τα συμφέροντα των 500 εκατομμυρίων των Ευρωπαίων που εκπροσωπούμε. Τίποτα δεν εμποδίζει τα κράτη-μέλη να συντονίζουν σε πραγματικού όρου την οικονομική του πολιτική. Είτε πρόκειται για το ιστορικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε πάνω απ' όλα την εξωτερική εκπροσώπηση τη Ένωση όπως πολύ σοφά μας είπε τώρα μόλις ο Ζων Κλοντ Γιούνκερ στα συμπεράσματά του. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Βολφ Κλίντς, φιλελεύθερη. Πέντε λεπτά. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Λυπούμε κι εγώ που είναι λίγοι οι συνάδελφοι σε αυτήν εδώ την πανηγυρική συνεδρίαση, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα ιστορικό γεγονός. Μιλήσαμε από τους ε, προλαλήσαντες πώς, ε, με πόση φυλακή με πόση επιφυλακτικότητα και δυσπιστία υποδέχθηκαν πολύ το ευρώ. Εάν όμως συλλογιστούμε πόσα διαφορετικά νομίσματα, χαρτονομίσματα, κέρματα αντικατέστησε και πόσους, α, φορεί χρηματοπιστωτικούς φορείς εκπροσωπεί και εκφράζει, θα μιλούσαμε μάλλον για Mission Impossible, για ε, μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Έχουμε να κάνουμε με ένα μικρό πολιτικό θαύμα έχουμε να κάνουμε με την υλοποίηση των υποσχέσεων του Βάλσταϊν του πρώτου ε, επιτρόπου ε, για την υλοποίηση αυτών των ε, οραμάτων για μια νομισματική πολιτική ενιαία. Έχουμε να ε, απαντήσουμε επίσης στους φόβους για τον υπερβολικό πληθωρισμό που θα προκαλούσε η εισαγωγή του ευρώ, ότι θα ανέβαιναν οι τιμές παντού. Απεδείχθη ότι ήταν ε, ψευδής αυτή η φόβη. Οι Ευρωπαίοι έχουν αποδεχθεί το ευρώ έχουμε να κάνουμε με ένα από τα λίγα σύμβολα που έχει στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός από τον ύμνο της και την Ευρωπαϊκή Σημαία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οικονομική πολιτική της Ευρώπης ε, δεν έχουν ακόμη βρει το ρόλο τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να αναπτύξει μια πολιτική σταθερότητας. Πρέπει πάντως να ε, σημειώσουμε για τα πρώτα 10 χρόνια του ευρώ ότι ο πληθαρισμός που παραμένει στα 2% σε εμάς, δηλαδή στο όριο του στόχους που είχαν προσδοριστεί, είναι σε σχέση με τα 50 χρόνια του γερμανικού μάρκου ε, πάρα πολύ επιτυχέ ποσοστό. Γιατί το Μάρκο, το οποίο θεωρούνταν υποδειγματικό νόμισμα προς τη σταθερότητά του, είχε πληθωρισμό 3%. Η ποιότητα όμως πάνω απ' όλα, η πραγματική ποιότητα του ευρώ αποδεικνύεται τώρα στην κρίση την οικονομική που γνωρίζουμε ότι παραμένει σταθερό, ότι είναι αποτελεσματικό, ότι πολύ γρήγορα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αποτελεσματικότητα αντιμετώπισε την κρίση και έδωσε σημάδια σταθερότητα και μηνύματα σταθερότητα όχι μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και προ τον έξω κόσμο. Και ταυτόχρονα είπε και πολύ σαφώ στι ΗΠΑ ότι επιτυχή οικονομική πολιτική μπορεί να έχει χωρί την εξάρτηση από την ιανδήποτε κυβέρνηση, αλλά ακριβώς χάρη στην ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας από την όποια κυβέρνηση, όποιες κυβερνήσεις. Τώρα τα κρατη μελη προχωρούν στην ανάπτυξη διαφόρων ε, προγραμμάτων συγκυρία για να αντιμετωπίσουν τι επιπτώσει και τη οικονομική κρίση στην ε, πραγματική ε, οικονομία. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται πάλι ενώπιον νέων προκλήσεων, γιατί εδώ διατρέχουμε τον κίνδυνο λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων ω προ την αντιμετώπιση αυτή τη κρίσεω, η σύγκληση που είχε μέχρι στιγμή επιτευχθεί εν μέρη μεταξύ των κρατών μελών τη ζώνη του ευρώ να απολεστεί. Έχουμε δηλαδή αυτό το κίνδυνο και πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε και όντως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης καλό θα είναι να μην ε, εξευτελιστεί. Αντιθέτως πρέπει να διατηρήσουμε την, ε, με αυστηρότητα τήρησή του όπως το παρελθόν και τώρα. Και πάλι θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια να παρακολουθεί την τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης από τα κράτη-μέλη με αυστηρή πειθαρχία. Ε, Επίση βλέπουμε ότι χρειάζεται στον χρηματοπιστωτικό τομέα να υπάρχει ένας ε, επόπτη, ένα ρόλο που θα μπορούσε να δραματίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή που θα μπορούσε να ανατεθεί σε μια κεντρική αρχή εποπτείας για τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί ο ρόλος του ευρώ, θα πρέπει τα κράτη της ζώνης του ευρώ να μιλούν με μία ενιαία φωνή και να εκπροσωπούμαστε στα νομισματικά και στον ΟΣΑ και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Παγκόσμια Τράπεζα με μία ψήφο με, έναν, ε, με μία ενιαία φωνή. Το να μιλούμε λοιπόν για μικροπράγματα ευτελίζει όλη αυτή την ε, προσπάθεια και την επιτυχία. Πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλούμε ενιαία, με ενιαία φωνή και έχουμε πολλές πιέσεις να αντιμετωπίσουμε και πολλά προβλήματα. Έχουμε τις μεγάλες δημογραφικές πιέσεις, έχουμε προβλήματα μεγάλα, έχουμε την παγκοσμιοποίηση ως ε, μεγάλο κίνδυνο και σε αυτό μπορούμε να απαντήσουμε με ως πρώτο βήμα βέβαια προς την κατεύθυνση αυτή τη της και της ενιαίας αντίδρασης των ε, ορισμό του Προέδρου της Ευρωζώνης αλλά ταυτόχρονα δεν αρκεί αυτό και πρέπει να προχωρήσουμε με άλλα αντίστοιχα μηνύματα. Η κυρία Μουσκαρδίνη παρακαλώ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά από δέκα χρόνια η αυξανόμενο, ο αυξανόμενος χώρος του ευρώ σαν νόμισμα και για τις διεθνείς συναλλαγές αλλά και για τα αποθεματικά δείχνει ότι το ευρώ είναι ένα διεθνές νόμισμα το οποίο συνεισέφερε στην οικονομική σταθερότητα και συνεισέφερε στις οικονομίες των χωρών που τη υιοθότησαν εκτός από οποιοδήποτε λάθος εκτίμηση τα οποία ενδεχόμενα ε, δημιούργησαν προβλήματα στους ε, πολίτες ε, γιατί ακριβώς όταν ε, ε, υιοθετήθηκε το ευρώ δεν έγιναν κάποια απαραίτητη έλεγχη. Το ευρώ υιοθετήθηκε χωρίς πολέμους, χωρίς ε, ηγεμονικές δραστηριότητες. Ήταν το αποτέλεσμα μιας ηθελημένης απόφασης που πήραν 11 κυβερνήσεις που πίστεψαν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση η οποία προβλέπεται από τις συνθήκες και συνεισφέρει στην δημιουργία αυτής της πολιτικής ένωσης η οποία ακόμα δεν έχει επιτευχθεί. Υπάρχουν κάποια προβλήματα προβλήματα, τα οποία όμως οφείλονται στην αποτελεσματικότητα ενός συστήματος, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί για να αντιμετωπίσουμε ένα άλλο στοιχείο, το οποίο είναι η εξέλιξη προς την, η ταχύτατη εξέλιξη προς την ε, ε, παγκοσμιότητα. Το ευρώ κλήθηκε να αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα, παραδείγματος χάρη αυτό της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και μας προστάτευσε από τις συνέπειες αυτής της διεθνούς κατάστασης. Αν δεν είχαμε το ευρώ θα επαναλαμβάναμε τις εμπειρίες του 1992. Σε αυτή την δέκατη επέτειο χαιρετίζουμε ε, την ε, είσοδο της, ε, στην Ευρωζώνη της, Σλοβα... Σλοβακίας. Και θεωρούμε ότι οι αποφάσεις και οι κινήσεις της Κομισιόν και της Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο. Όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες προσπάθειές μας, διότι δεν θα πρέπει η νομισματική πολιτική να απαγκιστρωθεί από την οικονομική. Σίγουρα η κατάσταση είναι ε, μοναδική. Έχουμε 11 κράτη με, την, ε, το νόμισμα, 27 κράτη τα οποία συντονίζουν την οικονομική τους πολιτική από την, ε, με, βάση αποφάσεις της Κομισιόν. Θα πρέπει να, ε, συντονίζουμε την νομισματική πολιτική με βάση μια κοινή οικονομική πολιτική η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως εάν οι οικονομικές αποφάσεις των κρατών μελών συντονιστούν από τις ε, κεντρικές τράπεζες ε, τις εθνικές και την ε, αιγίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας θα προχωρήσουμε. Αλλιώς θα έχουμε φοβερά προβλήματα διότι υπάρχουν και οι εξωτερικές προκλήσεις. Υπάρχει παγκοσμιοποίηση και αυτές είναι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι πρόσφατες εμπειρίες επιβεβαιώνουν την ανάγκη η Ευρώπη να, δει την, να αντιμετωπίσει την, τις αλλαγές. Θα πρέπει να υπάρχει πιο στενή σχέση ανάμεσα στις κεντρικές τράπεζες και στην, και στην Κεντρική Τράπεζα και τις, ε, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η πρόσφατη ενεργειακή κρίση απέδειξε ότι μια οικονομική, κοινή οικονομική πολιτική για τα βασικά στρατηγικά θέματα ή και τα θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες δεν θα πρέπει να καθυστερήσει, διότι η οικονομική πολιτική θα πρέπει να δημιουργηθεί και να στηριχθεί στο αυξανόμενο βάρος του ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των Κύριος Λίπιετς, για τρία λεπτά. Κυρίες και κύριοι. Κύριοι Επίτροποι, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω το ότι το 1992, τότε που η ψήφος της ε, Γαλλίας συνιστεί το όσον αφορά τη συνθήκη παρενέβη ο Ζακ Ντελόρ και είπε ότι και οι πράσινοι θα πρέπει να συμβάλλουν αυτό το 2% που έλειπε για να επιτευχθεί ο στόχος και είπαμε ότι μετά το ευρώ θα έχουμε την πολιτική Ευρώπη. Γιατί εάν έτσι δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε ο κόσμος ε, ποτέ δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια τέτοια πολιτική Ευρώπη. Όμως ε, το ευρώ έγινε, αλλά δεν ε, φτάσουμε στην πολιτική ολοκλήρωση της Ευρώπης και ακριβώς αυτό σήμερα μας απασχολεί. Το θέμα είναι γιατί θέλαμε τότε το ευρώ. Για δύο λόγους. Θεωρούσαμε ότι τα κριτήρια του Μαστρίχτ επρόκειτο να μας οδηγήσει σε κάποια κυκλική ύφεση για μια πενταετία τότε και επίσης ε, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να, ε, να αντισταθμίσουμε την ανεπάρκεια της συνθήκης του Μαστρίχτ όσον αφορά την ένταξη της νομισματικής πολιτικής στη γενικότερη πολιτική της Ένωσης και, σας το λέω ξεκάθαρα, ακόμα δεν με έχει πείσει η συνθήκη της ε, Μαστρίχτ, όμως όπως όλοι οι πράσινοι έχουμε πιστεί σε σχέση με τις ε, εξελίξεις που έχουν λάβει η χώρα και στην νομοθεσία αλλά και στην ε, πράξη όσον αφορά την ΟΝΕ και έχουμε τρεις βασικές αλλαγές που έχουμε δει πρώτα πρώτα η σταθερότητα τιμολογικής πολιτικής Έχουμε φτάσει στο 2% κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν είναι ε, ικανό σήμερα να αντιμετωπίσει ε, αυτήν την, ε, την κρίση που ταλανίζει τον κόσμο. Οι κινησιανές μέθοδοι δεν πιάσανε, οπότε αυτός ο στόχος του 2% πλέον δεν είναι αποτελεσματικός. Όμως, εάν δεν υπήρχε το 2% τότε θα είχαμε κάποια επιτόκια πραγματικά επιτόκια τα οποία δεν θα ήταν αυτό το οποίο επιθυμούσαμε, θα ήταν πολύ υψηλά. Επίση, έχουμε την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητα το 2005, ούτω ώστε σήμερα να μπορούμε να έχουμε μια πολιτική αποτελεσματική κατά τη κρίση. Άλλος μετασχηματισμό σημαντικός ήταν αυτός ο πάγιο διάλογος που γίνεται ε, Αλμούνια, Τρισέ, Γιούνκερ και Μπαρόσο αυτό είναι κάτι το οποίο αντιβαίνει ακόμα και στο γράμμα της νίκης του Μαστρίχτη γιατί αυτή η συνεργασία μεταξύ ας πούμε Τρισσό και Ελμούνια και από την άλλη μεριά Μπερνάγκη και Πόλσον ε, μας οδηγεί σε κάποια θετικά αποτελέσματα οπότε έτσι βλέπουμε κάποιες θετικές πλευρές της νίκης του Μαστρίχτη Αναφέρθηκαν οι προλαλήσαντες στην πολιτική των επιτοκίων, οπότε έτσι προσπαθεί το Συμβούλιο να καταλήξει σε κάποια επιτόκια, τα οποία να αντικατοπτρίζουν μια ρεαλιστική βιομηχανική πολιτική. Επίσης, ο στόχος της Κεντρικής Τράπεζας δεν είναι να έχει ένα επιτόκιο τόσο κοντά στο 2% αλλά να είναι κάτι το οποίο να δυστυχήσει και τη Λισαβόνα και να έχουμε επομένω μια πολιτική χρηματοδότηση του ιδιωτικού χρέους από την Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με Γκέτεπορ και Λισαβόνα. Επίσης, όπως είπαν προαλήσαντες, θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή υποπτία, κάτι το οποίο φυσικά γίνει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πρέπει να καλωσορίσουμε σε μερικά λεπτά τον πρόεδρο της Λετωνίας. Ε, θα πρέπει λοιπόν να εγκαταλείψω την έδρα για λίγη ώρα για να τον υποδεχθώ προσωπικώς όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Τώρα όμως συνεχίζουμε για λίγο. Η κυρία Φιγκεϊρέιντο για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με αυτή την ευκαιρία θα πρέπει να προβληματιστούμε βαθιά όσον αφορά τις συνέπειες της εφαρμογής αυτών των νεοφιλελευθερών πολιτικών σε σχέση με το ευρώ. Αυτές οι πολιτικές μας οδήγησαν στη σημερινή κρίση, σε ανισότητες, σε προβλήματα στην αγορά εργασίας, στην παινία. Προσοχή, να, πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Η σταθερότητα των τιμών δεν θα πρέπει να είναι μια πρόφαση, μια δικαιολογία για να προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποιήσεις και τα κράτη-μέλη να μην αναλάβουν τις ε, κοινωνικές τους ε, ευθύνες. Θα πρέπει να έχουμε κάποιες ελάχιστες ε, κοινωνικές εγγυήσεις, θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή μισθολογική πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχουν κολλήσει οι μισθοί, οι αυξήσεις είναι συμβολικές. Οπότε έχουμε οδηγηθεί σε πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις όπως συμβαίνει στη χώρα μου την Πορτογαλία. Έχουμε αυτό το καταστατικό αυτονομίας της τράπεζας. Αυτό όμως μας οδηγεί σε κάποια επιτόκια που οδηγούν εις υπερτίμηση του ευρώ, το οποίο δεν ωφελεί τους πιο αδύνατους, δεν ωφελεί τις πιο αδύνατες οικονομίες, δεν ωφελεί τις πιο αδύνατες ομάδες του πληθυσμού. Άρα όλη αυτή η πολιτική μας οδήγησε σε σύρρυγνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρέπει να πάμε τώρα σε μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων αναφοράς. Οι δε εργαζόμενοι, οι δε συνταξιούχοι, αυτή την δεκαετία βλέπουμε θέσεις τους να επιδεινώνεται. Οι δε ε, τράπεζες βλέπουν να αυξάνεται το ενεργητικό τους. Τώρα όμως έχουμε μια μεγάλη κρίση. και προσπαθούν με εθνικοποίηση να ιδιωτικοποιήσουν τα κέρδη τα οποία έχουν αποκομίσει στο παρελθόν. Όμως όλοι αυτοί, οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, όλοι αυτοί υποφέρουν από την κρίση. Και τα ωφέλη τους τελικά από τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται είναι πενταροδεκάρες. Προσοχή επομένως, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Προσοχή διότι σε ένα χρόνο διπλασίασαν τα κέρδη τους τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Γι' αυτό σας λέμε. Θα πρέπει να γίνει μια στροφή ριζική. Όχι στον οφειλελευθερισμό, όχι στον μονεταρισμό. Να σταματήσουν να ωφελούνται κάποιοι από τους φορολογικούς παραδείσους. Θα πρέπει και μέσω του κοινωνικού προπολογισμού να έχουμε πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου και να οδηγηθούμε σε κοινωνική συνοχή. Να μην έχουμε μία από τα ίδια. Και οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και ο σώζων είναι αυτόν Γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο θα οδηγηθούμε σε ακόμα χειρότερη κατάσταση και θα μεγαλώσει το χάσμα μεταξύ των οικονομιών της Ευρωζώνης. Να προστατεύσουμε τις ΜΜΕ και την παραγωγή τους είναι ποιοτική η παραγωγή τους. Να τους δοθούν κάποιες πιστώσεις. Και έτσι να προστατευτεί και η οικογένεια, να προστατευτεί η μεσαία τάξη, να έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και να καταπολεμήσουμε την παινία που ταλανίζει τόσο από τις χώρες μας. Ο Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρω ότι δεν έχετε τον χρόνο που φαίνεται εκεί, αλλά τέλος πάντων όταν χτυπάω το σφυράκι να ξέρετε ότι έχετε ολοκληρώσει το χρόνο σας. Ο κύριος Φαγάζα. Κυρίες και κύριοι, γιορτάζουμε την, τα 10 χρόνια του ευρώ, διότι είναι σαν να γιορτάζουμε τα 20 χρόνια. Εδώ αυτά που μου θύμισαν, αυτά που άκουσα εδώ, την Σοβιετική Ένωση στο παρελθόν. Όταν τα γιορτάζανε την επιτυχία των πενταετών προγραμμάτων πριν ακόμα ολοκληρωθούν με τους στόχους, με τα τρακτέρ, με τα στάρια που είχαν μαζέψει κτλ. Και ε, τι γίνεται, εδώ έχουμε ε, μία ερετούς Ευρωπαίους ηγέτες οι οποίες μας έδειξαν ε, πόσο ωραία πράγματα έχουν κάνει ενώ δεν έχει γίνει τίποτα. Πέρυσι τον Ιούλιο όταν η Ευρωπαϊκή τράπεζα, Κεντρική Τράπεζα ανέβασε τα επιτόκια όταν ε, διέλυαν, η αγορά και πέφταν τα επιτόκια. Αυτό είναι ένα σωστό θέμα το οποίο θα έπρεπε να θίξουμε. Αλλά αυτό δεν με εκπλήσει, διότι εδώ μιλάμε για μια πολιτική τάξη η οποία επιβάλλει τη θέλησή τους στις, ε, ε, στους Ευρωπαίους πολίτες. Μόνο η Δανία και η Σουηδία έκαναν ε, δημοψήφισμα για το ευρώ και αυτές το καταψήφισαν. Η ευρωζώνη δεν δοκιμάστηκε ποτέ. Τώρα θα δοκιμαστεί. Η Ισπανία είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Η Ιταλία και η Γερμανία λένε ότι δεν θα πρέπει ποτέ να μπουν στο, στο ευρώ. Για την Ελλάδα όμως η κατάσταση στην Ελλάδα ποια είναι. Χιλιάδες παιδιά βρίσκονται στο δρόμο και ε, διαμαρτύρονται και ζητούν από, τις κυβερνήσεις, από την κυβέρνησή τους να κάνει κάτι, να κόψει τη, τη, τα επιτόκια, να ε, υιοθετήσει μέτρα αποτελεσματικά για την ανάκαμψη της αγοράς. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα όμως η ελληνική κυβέρνηση, διότι είναι ε, δεμένη χειροπόδαρα από, την, ε, από, την, ε, από τις επιταγές ε, του ευρώ και θα πρέπει να περάσουν μέσα από την, ε, από την κάλπη. Εάν όμως δεν γίνουν εκλογές, η βία είναι η μόνη διέξοδος. Επομένως αυτό το οποίο κάνετε στην Ευρώπη είναι να κλείνετε τους ανθρώπους σε μια οικονομική φυλακή, σε ένα μπούνκερα. Και πώς θα βγουν από αυτό, θα χρειάζεται θάρρος, χρειάζεται ηγεσία και ενδεχόμενα χρειάζεται και αναπόφευκτη οικονομική ε, ε, ε, διάλυση. Όμως ξεχάστε, θυμηθείτε μάλλον ότι η, η Βρετανία που ήταν εκτός από το ευρώ μπόρεσε να υποτιμήσει, να κόψει τα επιτόκια, να κάνει πράγματα τα οποία έπρεπε να κάνει δεν ξέρω αν πήρατε είδηση ότι στην αγορά των ομολόγων τα βρετανικά ομόλογα ε, ε, έχουν πολύ σωστή ε, διαπραγμάτευση, διαπραγματική τιμή σε σχέση με τα γερμανικά επιτόκια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, αλλά καλό θα είναι να να, αν θέλετε να, να, κάνετε κάτι, δεν μπορείτε να αγνοήσετε την αγορά, δεν μπορείτε να, είσαστε, να, το, κάνετε, ε, να το παίζετε στουρθοκάμιλοι. Διότι εσείς μπορείτε να αγνοείτε, να αγνοείτε την αγορά, αλλά η αγορά δεν θα σας αγνοήσει. Enfin, dernier orateur... Τελευταίος ομιλητής για τη συζήτηση αυτή. Και θα τον ακούσουμε με ησυχία, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Έλμερ Τρία λεπτά. Πρόεδρε, τα τελευταία 200 χρόνια τουλάχιστον 5-6 προσπάθειες έγιναν για ενοποίηση νομισματών ή τουλάχιστον νομισματικών μηχανισμών, ισοτιμιών και απέτυχαν ικτρά εις βάρος των συμμετεχόντων. Το ίδιο συμβαίνει και με το ευρώ. Οι ανισορροπίες που είχαν προβλέψει οι επιφυλακτικοί, οι επικριτές του ευρώ αποδεικνύονται ήδη. Η Ιταλία ε, έχει καταρρεύσει. Η Ισπανία ξεκινάει σε μια ταυρομαχία με μεγάλη ορμή και ε, δόξα και καταραίει μέσα στο αίμα και, τη σκόνη. Η Ελλάδα καταραίει υπό το βάρος ενός υπερτιμημένου ευρώ. Η ισοτιμία ομολόγων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας έχει φτάσει σε σημείο ε, κατάρρευσης πάνω από 200 μονάδες. Δηλαδή εμείς στη Βρετανία έχουμε προστατεύσει το δικό μας νόμισμα και δεν κινδυνεύουμε από το τεστραμένο τρένο του ευρώ, του ευρώ το οποίο βαίνει αργά και σταθερά προς τον κρέμο. Χρόνια σας πολλά για το ευρώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και τώρα προχωρούμε στις ψηφοφορίες.